Uh, Αγαπητοί συναδελφοί, τώρα τα μηχανήματα δουλεύουν πια, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε. Σας καλωσορίζω όλους και σας ενημερώνω ότι όσο ήθιστε η συνεδρίαση αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Αρχίζουμε με το σημείο 1 στην ημερήσια διάταξη που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. 21 Σεπτεμβρίου σας μοιράστηκε. Δεν άκουσα τίποτα αντιρρήσεις. Έχετε τώρα μήπως καμιά πρόταση για αλλαγή, παρατηρήσεις, όχι. Ωραία, τότε θεωρείται εγκεκριμένη. Σημείο 2. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσει. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη που είναι η ψηφοφορία. Για την ψηφοφορία θέλω να σας δείσω πρώτα να κάνουμε μια δοκιμή για τις κάρτες σας. Για βάλτε τις κάρτες στο μηχάνημα παρακαλώ. 21 κάρτες, 22 έχουν μπει στο μηχάνημα μέχρι τώρα. Άρα χρειάζονται και άλλοι για να φτάσουμε στους 25. So not everybody just... Δεν ψήφισατε όλοι, εγώ για παράδειγμα. Αλλά δουλεύει το δικό μου το μηχάνημα. Αρχίσουμε με την πρώτη λοιπόν ψηφοφορία που είναι η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μεγάλη ψηφοφορία αυτή. Αρχίσουμε με τη συμβαστική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190 υπέρ. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 120. Συμβαστική. Συμβαστική 2. Υπέρ. 2. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 131 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 133. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 11, 134 τώρα υπέρ. Του L. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 136. «136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ, 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 149 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει και η 150, 152 152 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 162 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 162 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 Α, συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 170, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίας απορρίφθηκε. 5-18. 171 τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 180. Ψηφίστε παρακαλώ. FTT παραπάνω. Όχι. Α. Λοιπόν, ένας από το FTT και ένας από το NF πρέπει να μην ψηφίζουν στην ψηφοφορία γιατί το μηχάνημα αντιδρά. Λέει ότι έχουμε ένα παραπάνω από την κάθε ομάδα. Τι, σφάλει το μηχάνημα, είσαστε σίγουρος. Μόνο εσείς ψηφίζετε λέτε. Και από το EFDD. Ωραία, άρα να ελέγξουμε τα μηχανήματα. Ξανά, ξανά. Για την 180 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Για να δούμε πάλι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει πρόεδρος. Αλλά πρέπει να το κοιτάξουμε. Αλλιώς θα πρέπει να ψηφίζουμε κάθε φορά δυνατά στο σκυρός, ε. Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό.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 don't want to then be accused that there was something wrong with Maybe the vote. changing machine, I don't know. Change machine. Yeah, could, could we ask the two... Παρακαλώ τους δύο συναδέρφους, μήπως θα μπορούσατε να αλλάξετε θέση, να πάτε σε κάποιο άλλο μηχάνημα, μήπως κάτι αλλάξει, μήπως φταίνε τα μηχανήματα που ήσασταν. Αλλάξτε θέση λοιπόν. Και τώρα Ξανά κάνουμε τη δοκιμή. Το ίδιο. Το ίδιο. Άρα κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα, ε. Φοβερό. It's not true. We can take... Yeah. the colleagues, there will be, I mean, we, we probably can... Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα θα είναι με την ονομαστική ψηφοφορία. No, because nobody is voting. Could we start voting Για να ψηφίσουμε πάλι, γιατί έχουμε τον τεχνικό τώρα μαζί μας. Βλέπετε, αμέσως εμφανίζεται σαν παραπάνω.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 ελέγχαμε έτσι κι Αλλιώ θα πάμε διανατάσσεω τη χειρός. Λοιπόν, στο μεταξύ, διανατάσσεω τη χειρός, δεν έχουμε άλλη επιλογή. 180, υπέρ παρακαλώ. 180. Μετράμε. Κατά. Αποχές. Τώρα πρέπει να είναι εντάξει, λέει ο τεχνικός. Τώρα είναι εντάξει τα μηχανήματα. Οπότε 180 με το μηχάνημα. Ψηφίζουμε για την 180 ηλεκτρονικά. Μα τώρα δεν δουλεύει καθόλου, λέει ο πρόεδρος. Τώρα είναι το ΕΛΚ που έχει έναν παραπάνω. Εντάξει, δεν ψηφίζετε εσείς. Καλώς. Ψηφίζουμε για την 180, ε. Και μην αλλάξετε γνώμη. Μπορεί να είναι βαρετό, αλλά ψηφίστε το ίδιο, παρακαλώ. Τώρα έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα είναι εντάξει, κρατήστε την κάρτα σας με την έχετε στο μηχάνημα. Λοιπόν, 180 τελευταία ευκαιρία να ψηφίσετε για την 180 ηλεκτρονικά. Ε, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 196 υπέρ, 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω η 199 αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Δεν λειτουργεί. Δεν ψηφίζετε όλοι όμως συνάδελφοι. Πέρα της φοφορίας απορρίφθηκε. 200 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 200... Α, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά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 απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για τη 18 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Α, ξανά. Ψηφίστε.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 Μα δεν ψηφίζετε, θα ελέγξουμε. Αφού δεν σηκώνετε τα χέρια καλά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε μια προφορική τροπολογία στην 30. Αντιτίθεται κανείς? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν με την προφορική τροποποίηση. 30 ε, λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 κατά πίπτη, 32 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 40 υπέρ, κατά απορρίπτεται 41 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 54. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας απορρίφθηκε. 55 έχει αποσυρθεί, 56 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε την 57. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφορίας απορρίφθηκε. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε 61 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Νομίζω, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την 61. Ψηφίστε παρακαλώ. Πάλι κάποιο λάθος έγινε. Ωραία, ψηφίζουμε τώρα για την 61 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίζουμε για την 61 ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, 64. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρασε τη φοφορίες. Απορρίφθηκε. 65 υπέρ κατά αποχές 65 υπέρ κατά α, απορρίφθηκε αλλά όχι, θα ελέγξουμε καλύτερα για να είμαστε σίγουροι νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά σας βλέπω αναποφάσεις τους πέρα στις φοφορίες Απορρίφθηκε. 9-11 το αποτέλεσμα. 66 τώρα. Υπέρ. Κατά. Το ίδιο. Θα ελέγξουμε και για την 66 λοιπόν. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρασε της προφορίας. Απορρίφθηκε. 67 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. 77. Εντάξει, θα ελέγξουμε πρώτο τμήμα της 77 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Μάλιστα, δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Χωρίς αμφιβολία. 78, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας. 79 τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές κανείς δεν ψηφίζει. Αυτή είναι η ελευθερία ψήφου. 81. Παρ' όλα αυτά, ηλεκτρονικά, παρακαλώ, να ελέγξουμε για την 81. Ψηφίστε. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 84 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87 αποσύρθηκε. 88 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της 90 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 99 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. 100 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σηκώνεται χέρια. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 103. Πέρασε τη εγκρίθηκε. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 106. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίας. Εγκρίθηκε. 11-10. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Από... Ε, δεν σηκώνετε τα χέρια σας εσείς εδώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Από το ΕΛΚ. Α, 109. Πέρα τη ψηφοφορια απορριφθηκε Απορρίφθηκε 10-10 ισοψηφία. 219 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 223 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αποσύρθηκε 225, τροπολογία 1 υπέρ. Α, δεν την αποσύρεται. Τότε ψηφίζουμε τη 225. Δεν μπορώ να έχω ονομαστική ψηφοφορία όμως. 225 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Ε. Δεν είμαστε σίγουροι. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη 225. Μπορείτε να ψηφίσετε. Κάποιος δεν ψηφίζει. Τι να κάνουμε. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. 226 τώρα. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Η καταπίπτει. Το δεύτερο ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος 226. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε δεύτερο τμήμα του 226 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην 227 υπέρ. Το έλκο δεν το γνωρίζει νομίζω. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Συμβαστική 9 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 256 χωριστή ψηφοφορία. Πέρας πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για το τρίτο μέρος υπάρχει η προφορική τροπολογία. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος της 256 πέρα. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Τρεις δεν ψηφίζουν, δεν θέλει να ψηφίσουν. Τι να κάνουμε. Πέρας. Α, τώρα μου ψηφίσατε. Λοιπόν, απορρίπτεται. Παίρναμε στο τρίτο. Α, ε, στην προφορική τροπολογία επί του πρώτου μέρους. Να αντικαταστήσει το πριν από τη μέρα των εκλογών μέχρι πριν από την πρώτη μέρα των εκλογών. Υπέρ. Κατά. Αποχές τεκτό. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την συμβιβαστική 10 γιατί δεν ψηφίσατε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και γίνεται δεκτή. Δεκτή λοιπόν η 10. Συμβιβαστική 11 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται δεύτερο μέρος περ, κατά. Να το επαληθεύσουμε. Το δεύτερο μέρος της 11. Πέρας. Δεκτή. 2.38 Μέρος πρώτο Υπέρ Κατά Αποχές απορρίπτεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές για να δω να το επαληθεύσουμε με συγχωρείτε άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινείται η 2-3 πίπτη. Λοιπόν, 2 2-39 υπέρ. Κατά. Ε, 2-41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.45 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά εποχές δεκτή 2.49 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.50 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 2.51 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε τη 2.51 Πέρας. Δεκτή. 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 προφορική ποιος είναι κατά κατνής οπότε την ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 2.55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.57 προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά να την επαληθεύσουμε. Είναι ίδια. Όχι, ψηφίσαμε. Την ψηφίζουμε, τι κάνουμε. 2.57 ε, ψηφίσμα τελικά. Άρχιδη η ψηφοφορία. Γιατί δεν κατάλαβα τι μου λέγατε με το σώμα. Απορρίπτεται λοιπόν ελαφρώς. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.59 υπέρ. Α, α, μάλιστα, συγγνώμη. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2.64 υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι είναι δεκτό. 2.64 λοιπόν να το επαληθεύσουμε. 2.64 άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία, πέρας και γίνεται δεκτή. 2.65 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.66 ε, καταπίπτει. 2.67 καταπίπτει. 11. Την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. 269 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 273 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται 2.74 υπέρ κατά εποχές ε, απορρίπτεται 2.84 προφορική τροπολογία 2.84 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά να το δούμε απορρίπτεται 2.75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.81 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Υπάρχουν τεχνικές ε, τροπολογίες για την ορολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τώρα, τελική ψηφοφορία. Πρέπει να διαβάσω τα πράγματα λοιπόν. Που τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης που περιλαμβάνει και εντολή για αλλαγή του νόμου του 1976 για να διαβιβαστούν στο Συμβούλιο. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Τζορτζ, τι, επειδή δεν το ξέχασες, τι γίνεται. Α, απλά, λέω μήπως. Πέρας και βεβαίως εγκρίνεται 14 υπέρ 5 κατά 3 αποχές. Περνάμε τώρα σε Στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Ψηφίζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Hello.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 ε, συγγνώμη δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω, κάνω δύο χέρια. Λοιπόν, υπέρ, πέτει ένα, υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε γιατί δεν είναι σαφές. Εγκρίνεται λοιπόν. Γιούρι ένα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές δεκτή Ευχαριστώ χωριστή ψηφοφορία για την ΔΕΛΤΑ. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές ε, κατά ε, δεκτό, ε, τρίτο μέρος πέρα, κατά. Να, ξαναψηφίζουμε για το τρίτο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Δεκτή. Λοιπόν, συμβαστική ε υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Γιούρι 3 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή συμβαστική F υπέρ κατά αποχές δεκτή Γιούρι 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή Γιούρι 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική G υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά να την επαληθεύσουμε άρχεται την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή συμβαστική H η 40 πέρασε μόνο εσείς ήσασταν κατά να την επαληθεύσουμε αν θέλετε θέλετε να επαληθεύσουμε ωραία να επαληθεύσουμε την τροπολογία 40 άρχεται η ψηφοφορία 40 άρχεται η ψηφοφορία άλλος ένας για να κλείσει ωραία εγκρίνεται λοιπόν συμβαστική H υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Πέτη 13 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Ναι, ναι, το ίδιο. Συμβαστική Άι υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Γιούρι 5 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική W υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ψηφίζουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία Πέρας και απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την 48 με προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας, όχι. Την ψηφίζουμε. 48 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. J υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. Συμβιβαστική K υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές δεκτή 5-9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική M υπέρ κατά αποχές δεκτή Γιούρι 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 ε, υπέρ 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πέτει 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε νομίζω. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέτει 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5-16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5-17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική π. Όχι. Όχι, π. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Q. Όχι, εδώ κάνω λάθος. Ή, κάνω, ή δεν κάνω δεν κάνω, γιατί έχει αποσύρθει 79 υπέρ της συμβαστικής κατά αποχές εγκρίνεται, 83 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 5. 8. Ψήφι υπέρ. Έχει ζητηθεί τμηματική ψηφοφορία. Ναι. Πράγματι, για την ΑΡ είχε ζητηθεί τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 5 8, ψήφι υπέρ Ναι, είναι δύσκολο να καταλάβω από τα χρώματα. Σίλβι, θέλατε κάτι να πειτε Πέτη οκτώ ψηφίζουμε. Υπέρ. Υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την οκτώ της Επιτροπής Αναφορών. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική S, υπέρ, είναι τμηματική, μάλιστα. Πρώτο τμήμα της S, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να πάμε στην... Ορίστε. 22 in favor. 22 πέτη υπέρ, κατά. Κατά. Δεν ψήφισαν οι του ΕΛΚ. Υποθέτω ότι είναι κατά. Απορρίπτεται. Α, απορρίπτεται μάλιστα. Ωραία. Πάμε στη συμβαστική. Τι τμήματα. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέτει 26 ψηφίτε κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 15 υπέρ κατά ελέγχουμε τη Γιούρι 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται 10 προς 11. Συμβιβαστική Γιού σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Α, έχουμε, έχουμε κάποιες άλλες τροπολογίες που προηγούνται. 109 τροπολογίες, το συγγνώμη. Απλά πρέπει να μου μιλάει ένας, όχι και δύο ταυτόχρονα. 109 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά. Αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμφωνείτε. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 110. Πέρασε. Απορρίπτεται 10 προς 11. Προπολογία 111 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 111. Πέρασε τις Αυτή τη φορά ανάποδα, 11 προς 10, εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβιβαστική U. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, να ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, Ξέρετε, σε περιπτώσεις στην Ολομέλεια έχει τύχει να έχουμε 9 τμήματα ή 11. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Πρέπει να το ελέγξουμε όμως. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της γιου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πού πάμε τώρα. Στην τροπολογία 119. Ψήφι υπέρ. 11 προς 9 ήταν το προηγούμενο αποτέλεσμα. Πραγματικά είμαστε διαρρεμένοι, πολύ κοντά. Τροπολογία 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 τροπολογία. Ψήφι περ 123. περ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, δεν ξέρω. Πέρας φοφορίας. Εγκρίνεται. Γιούρι 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 3 υπέρ. Κατά. Υπέρ ξαναλέω. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτη 10 Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω. Ο μόνος που ψηφίζει είναι ο Τζόρτς από την ομάδα του ΕΛΚ. Δεν ξέρω και αν σας ακολουθούν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λέω να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 5-10. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πέτη 24 υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Αποχές δεν εγκρίνεται. Γιούρι 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά Άποχες απορρίπτεται. Πάμε τολική σκέψη και αναφορές. Ε, τροπολογία 1 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Πρώτο τμήμα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές από Ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ακούω κάτι φωνές και δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Τέλος πάντων, ε, τμήμα 2 υπέρ. Δεν έχει νόημα βέβαια. Sorry, just somebody who works on the compromises could, uh, could... Να μας εξηγήσει κάποιος που έχει καταλάβει τι γίνεται με τις συμβαστικές. Νομίζω ότι αν απορρίψουμε ένα κείμενο χωρίς κάποιες λέξεις, δεν έχει νόημα μετά να ψηφίζουμε τις λέξεις, αφού ψηφίσαμε το κείμενο χωρίς, δηλαδή το τμήμα χωρίς τις λέξεις. Κύριε Σέφλιν, ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι έχουμε τη λύση στο πρόβλημα. Είμαστε στην Α που έχουμε τρία τμήματα. Το πρώτο χωρίς κάποιες λέξεις και ακολουθούν τα άλλα τμήματα με κάποιες από αυτές τις λέξεις. Καταψηφίσαμε το πρώτο τμήμα. Σέπφλιν. Σύγνω στον κατάλογο ψηφοφορίας υπάρχει ένα λάθος. Έπρεπε να είναι θετικό το, το πρόσημο στο πρώτο τμήμα, ενώ εδώ έχει μείο, έχει πλήν. Επιτροπή, συμφωνώ να ξαναψηφίσουμε, γιατί υπήρξε παρανόηση, να, καταψη, να, ξαναψηφίσουμε το πρώτο τμήμα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Άρα να ξαναψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της συμβαστικής α. Πρώτο τμήμα λοιπόν. Ξαναψηφίζουμε. Το ΕΛΚ τώρα πρέπει να είναι υπέρ. Υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην Η συμβαστική W έχει απορριφθεί, άρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 8. Κατά. Επαναλαμβάνω, ψηφίζουμε την τροπολογία 8. Είχαμε τη συμβαστική W που απορρίφθηκε έξω και πρέπει να ψηφίσουμε την 8. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές πάλι απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική B υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ανακαλύψαμε ότι επειδή απορρίφθηκε η W, Η συμβιβαστική, θα πρέπει να ψηφίσουμε και την τροπολογία 58. Πάτε πίσω παρακαλώ λοιπόν στην 58, σελίδα 8. Είναι πριν τη συμβιβαστική L, ακριβώς από πάνω έχει την τροπολογία 58. καλύπτω το W, αλλά αυτή απορρίφθηκε. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε και την 58 τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά μπορούμε να το ελέγξουμε. Γιατί δεν σκόφηκαν και πολλά χέρια. Τροπολογία 58, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το σύνολο της έκθεσης ονομαστικά. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Ομόφωνα. Ομόφωνα εγκρίνεται. Τζορτ δεν είναι για λόγο εσού, αλλά για τους πολίτες. Και εγώ πολίτης είμαι. Συγχαρητήρια, Τζόρτζ. Περνάμε τώρα στην τρίτη για σήμερα ψηφοφορία που ελπίζω και εδώ να έχουμε την ίδια θετική έκβαση. E Πρόκειται για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών.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 Ψηφίσουμε τώρα όμω για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα Ηνωμένα Έθνη. Έχουμε τη συμβιβαστική Α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβαστική ΣΥΓΑΜΑ. γάμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ Εκτός μικροφώνου παρέμβαση, δεν την ακούμε. Η 12 καλύπτεται, λέει η πρόεδρος, αλλά μπορεί να έχω αν λάθος. Καλύπτεται όμως. Λοιπόν, είμαστε συμβαστική γάμα υπέρ. Α, ψηφίσαμε. 15, τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D, δέλτα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ή. Υπάρχει μια κατατμήματα ψηφοφορία εδώ. Ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το πρώτο τμήμα της συμβιβαστικής ε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα τώρα της συμβαστικής ε υπέρ κατά ίδια πλειοψηφία νομίζω θα ελέγξουμε καλού κακού ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής ε. Θα ελέγξουμε. Δεν βλέπω να ψηφίζετε όλοι. Πέρα της οφορίας Απορρίφθηκε. 9-11. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 24. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 24 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 10-11. 25. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά πάμε στην 27. Υπέρ παρακαλώ. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Αντιτίθεται κανεί. Όχι. Ωραία. Υπέρ παρακαλώ του 27. Κατά. Ψηφίστε. Ηλεκτρονικά να ελέγξουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 19. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και εδώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τις ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 30 υπέρ. Θα ελέγξουμε γιατί και εδώ βλέπω τσίμα τσίμα το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της οφορίας εγκριθηκε 11.8. Τροπολογία 32 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίφθηκε. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 35. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίες. εγκρίθηκε. 36 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 38 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρα στις οφορίες 11-10 εγκρίνεται. 39 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται έτσι. Καλά, να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για την 40 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 41. Έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα τη 41 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Ο Ποιο είναι, ο Βίλαντ είναι που το λέει. Στην Ολομέλεια, μην τραβάτε τις κάρτες σας από το μηχάνημα πολύ νωρίς, γιατί δεν καταμετράτε η ψήφος τότε. Και είναι ονομαστική ψηφοφορία εδώ, οπότε να, η κυρία που έφυγε πριν και έβγαλε γρήγορα την κάρτα από το μηχάνημα, δεν καταμετρήθηκε η ψήφος της. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Γκίθερ Χόφστατ θα μας παρουσιάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη διογρανική συμφωνία για την βελτίωση της νομοθεσίας. Είναι στο δρόμο. Οπότε θα περάσουμε σε αυτό το σημείο που είναι το τελευταίο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα πολύ σύντομα. Όσοι θέλετε να ακούσετε τον κύριο Φερχόφστατ και να έχετε ανταλλαγή απόψεων, μαζί του μη φύγετε από την αίθουσα.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

like to start this part of... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο τμήμα της συνεδρίασής μας, οπότε όσοι επιθυμούν να παραμείνουν, καλώς. Θα δώσω το λόγο στον Γκίφερ Χόφστατ, ο οποίος ε, συμφώνησε να έρθει σήμερα εδώ και να μας παρουσιάσει την πορεία των ε, διαπραγματεύσεων σχετικά με την Διοργανική Συμφωνία για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, μια που είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γκί, Θέλεις να υπενθυμίσεις τους συναδέρφους πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν τον Ιούνιο, έτσι δεν εκεί. Συμμετέχουν δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η δικιά μας που είναι αρμόδια για τις διοργανικές σχέσεις. Όταν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις και συμφωνήσουμε πάνω σε κείμενο, εμείς έχουμε την ευθύνη να πάμε την έκθεση στην Ολομέλεια για να την ε, εγκρίνει. Γι' αυτό και έπρεπε να συμμετέχουμε. Και γι' αυτό έχουμε υποβάλει και τις θέσεις μας γραπτά πριν το καλοκαίρι. Ε, δεν ξέρω είναι σωστό να πω ότι είμαστε τυχεροί, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα είναι πολύ καλό που μέλος της Επιτροπής μας, ο Κίφερ το ορίστηκε ως ο ε, αρμόδιος, ως εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως υπεύθυνο δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις διαπραγματεύσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξω απόψεις μαζί σας για τις διαπραγματεύσεις αυτές σχετικά με τη Διοργανική Συμφωνία για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας. Όπως είπατε ήδη, ορίστηκα διαπραγματευτής από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο. Οι συζητήσεις μεταξύ των τριών οργάνων άρχισαν αμέσως μετά τις θερινές διακοπές. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι έχει επιτευχθεί στο μεταξύ κάποια πρόοδος. Βασικά οργανώνουμε τη δουλειά μας σε δύο ομάδες. Έχουμε μια τεχνική ομάδα με υψηλού επίπεδου υπαλλήλου που κάνουν προτάσεις και υπάρχει και μια ομάδα σε πολιτικό επίπεδο η οποία παρτίζεται από τον ε, Υπουργό Σμιτ από πλευρά τη Προεδρία, τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εμένα τον ίδιο. Και εμεί εξετάζουμε τα προτινόμενα κείμενα. Δύο συναντήσει είχε μέχρι τώρα η ομάδα πολιτικού επίπεδου και μία τρίτη θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η τρίτη συνάντηση δηλαδή που οργανώνουμε. Το κλίμα στις συναντήσεις αυτές είναι εξαίρετο. Και η Λουξεμβουργιανή Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ε, δείξει την πραγματική τους πρόθεση για να πετύχουμε αποτελέσματα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αυτές και στόχος κοινό και των τριών είναι να ολοκληρώσουμε πριν από τα τέλη της χρονιάς αυτής ή δυνατόν οργανώνουμε ως εξή τις συναντήσεις μας και τις συζητήσεις. Αρχίσαμε και θα επανέλθω σε αυτό με τον προγραμματισμό που είναι το κεφάλαιο αριθμός 2 μιας πιθανής συμφωνίας. Τώρα συζητάμε για τα μέσα που θα μας βελτιώσουν την νομοθεσία. Ε, διαβουλεύσεις, εξ post, ε, αξιολογήσεις κτλ. Αυτό είναι το κεφάλαιο 3. Και συμφωνήσαμε επίσης για το ότι εκτός από την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα υποβάλουν συγκεκριμένα κείμενα όσον αφορά τα υπόλοιπα κεφάλαια της συμφωνίας αυτής. Τώρα επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω λιγάκι την ουσία του έργου μας, τι έχουμε κάνει ακριβώς μέχρι τώρα και ποιες είναι οι προοπτικές που μας περιμένουν στα επόμενα βήματά μας. Και το κεφάλαιο 2 πρώτα απ' όλα που είναι ο προγραμματισμός. Εδώ συμφωνήσαμε ε, καταρχήν επί ενός κειμένου όσον αφορά τον προγραμματισμό. Αλλά όπως γνωρίζετε ο βασικός κανόνας στην πολιτική είναι ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα. Συνεπώς, θα μπορούμε να σας δώσουμε ένα τελικό κείμενο μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί διαπραγματεύσεις και έχει συμφωνηθεί ολόκληρο το κείμενο. Αλλά αν θέλετε μπορώ να σας ενημερώσω για το περιεχόμενο αυτού του πρώτου κεφαλαίου το οποίο ολοκληρώσαμε, που είναι ο προγραμματισμός όπως είπα. Προσπαθήσαμε να έχουμε καλή ισορροπία συνένεση και των τριών πλευρών, αλλά συγχρόνω φροντίζουμε να διασφαλίζουμε τα συμφέροντά μας, εκείνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και θα αναφέρονται και ο πολιετής προγραμματισμός και ο ετήσιος προγραμματισμός και τα δύο. Για τον πολιετή προγραμματισμό εκεί θα υπάρχουν πολιτικοί στόχοι για πέντε χρόνια, ενώ ο ετήσιος προγραμματισμός θα καθορίζει προτεραιότητες για την επόμενη κάθε φορά χρονιά. Θα υπάρχουν και διατάξεις επί του περιεχομένου του Προγράμματος Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία κλειδί εκείνα πάνω στα οποία θέλουμε να συμφωνήσουμε για έναν πολιετή προγραμματισμό αλλά και ποιες είναι και οι υποχρεώσεις ε, τι μπορεί να αποσυρθεί ή τι μπορεί επιπλέον να ζητηθεί ως πρόταση από τους άλλους νομοθέτες. Όταν μιλάμε λοιπόν για προγραμματισμό, εδώ δεν πρόκειται μόνο για το περιεχόμενο του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν, πρόκειται και για την αντίδραση από τις άλλες πλευρές. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε θα ζητήσει να αποσύρει κάποια νομοθετική πρόταση ή αντίθετα να προσθέσει μια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί έτσι δεν πρόκειται, όπως λέω, μόνο για το περιεχόμενο, αλλά πρόκειται και για τις αλλαγές στις νομοθετικές προτάσεις, είτε αυτές αποσύρονται είτε προτείνονται νέες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάναμε και μια χειρονομία προς το Συμβούλιο. Πολλά βέβαια εκείνοι μας χρωστούν σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Δεχτήκαμε ότι σημερι... όπως υπάρχουν διμερείς συζητήσεις Επιτροπής και Κοινοβουλίου, θα μπορούν να υπάρχουν και διμερείς συζητήσεις Επιτροπής και Συμβουλίου επί του προγράμματος εργασίας της Κομισιόν. Αλλά πρέπει να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Διασφαλίσαμε σε αυτή τη χειρονομία, σε αυτή τη συμφωνία, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε επιτρέπει, ούτε θα συμφωνήσει ποτέ με αποδυνάμωση του προηγούμενου πλαισίου του 2010. Ξέρετε ότι συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο τότε δεν ενδιαφερόταν για συμμετοχή, αλλά έκτοτε μετά τη συμφωνία αυτή του 2010 το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι μια τέτοια συμφωνία ανάμεσα στο εκτελεστικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νομοθετικό είναι κάτι που δεν φτάνει. Οπότε, στο τέλος, στη συμφωνία, δεν θα υπάρχει κείμενο ή άρθρο το οποίο να μειώνει τις φιλοδοξίες ή το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας του 2010 όσον αφορά την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ό,τι υπήρχε, υπάρχει, οι φιλοδοξίες εκείνες δεν είναι δυνατόν να μειωθούν με αυτή τη νέα συμφωνία για τις διμερείς επαφές Συμβουλίου Κομισιών. Αυτό όσον αφορά τον προγραμματισμό. Ε, υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες, βέβαια και το Κοινοβούλιο δεν είναι λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν. Γιατί στα μέσα του προγραμματισμού αυτού έχουμε και την κατάσταση πραγμάτων στην Ένωση, που είναι σημείο κλειδί όπου το περιεχόμενο του προγραμματισμού, του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτεται. Μπορεί να το κάνει και στο Συμβούλιο. Αυτό δείχνει ότι μπαίνουμε σε ένα κανονικό ε, σύστημα όπου έχουμε το εκτελεστικό βραχίωνα, την Κομισιόν και στη συνέχεια δύο νομοθετικούς που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης και το Συμβούλιο που εκπροσωπεί τις χώρες μέλη. Αυτά περί προγραμματισμού. Η επόμενη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα αρχίσει με τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ένα δύσκολο ζήτημα είτε πρόκειται για διαβουλεύσεις, είτε πρόκειται για εξπόστ αξιολογήσεις. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η συζήτηση αυτή. Η Κομισιόν έχει κάποιες προτάσεις που εμείς μέχρι τώρα ως Κοινοβούλιο θεωρούμε παράδεκτες, αλλά η Κομισιόν θεωρεί ότι εφόσον υπάρχει νέα συμφωνία δεν μπορεί να μείνει σε ένα status quo, γιατί τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε για βελτίωση της νομοθεσίας. Εγώ δεν συμφωνώ ακριβώς και γιατί, γιατί οι αξιολογήσει αντικτύπου για παράδειγμα είναι ένα μέσον το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί για να βοηθηθούν στις αποφάσεις που παίρνουν. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο και δεν εμποδίζει τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαδικασία, τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων. Υπό το φως λοιπόν της εντολής υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής. Την επόμενη φορά ελπίζω να έχουμε μια συμφωνία βέβαια με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αλλά ποιες είναι οι δυσκολίες. Η υποχρέωση των νομοθετών να κάνουν μελέτη αντικτύπου για τις δικές τους τροπολογίες. Εμείς λέμε ότι δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο γιατί αυτό περιορίζει τη νομοθετική εξουσία του σώματος εφόσον μπει ως προϋπόθεση. Δεύτερον, η Κομισιόν προτείνει ένα ανεξάρτητο πάνελ το οποίο να μπορεί να εξετάζει τις τροπολογίες της ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της όποιας πρότασης της Κομισιόν. Και αυτό λέμε εμείς ότι είναι μια επιπλέον δυσκολία. Και το τρίτο είναι η διαβούλευση των διαφορεμένων μερών από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προηγουμένω έχει εγκρίνει την πρότασή τη. Οχτώ εβδομάδε, δηλαδή μετά την προθεσμία που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό είναι προβληματικό για μα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πολύ προτιμότερο οι διαβουλεύσεις να λαμβάνουν χώρα πριν εγκρίνει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν το καταλαβαίνω αλλιώ. Συνήθω πρώτα διαβουλεύεσαι και μετά κάνει μια πρόταση. Δεν είναι δυνατόν πρώτα να κάνει την πρόταση και μετά να έχει διαβούλευση. Ελπίζω να το κατανοήσουμε τέλο πάντων στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων το γιατί βάζουν τα άλογα πίσω από το κάρο αντί μπροστά από το κάρο. Όπως λέμε στα γαλλικά. Λέει ο κ. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι οι διαβουλεύσεις πρέπει να λαμβάνουν χώρα πριν υποβληθεί η πρόταση και τι πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να αρχίζει κάθε νομοθετική διαδικασία και όχι ανάποδα. Αλλιώς μπερδεύει στην νομοθετική διαδικασία τους ενδιαφερομένους. Είναι το αντίθετο από αυτό που ήθιστε. Στις χώρες μας. Κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με νομοθετική διαδικασία. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία εμπόδια. Τα τρία ζητήματα. Ναι λοιπόν υπάρχει μελέτη αντικτύπου αλλά τότε πρέπει να είμαστε εμεί υπεύθυνοι. Και δεν μπορεί μια τέτοια διαδικασία να εμποδίζει την νομοθέτηση. Επίσης, διαβούλευση ναι, αλλά πριν γίνει η πρόταση και όχι μετά. Παρά λοιπόν τις τρεις αυτές διαφωνίες που έχουμε, και το Συμβούλιο εδώ συμφωνεί μαζί μας, έτσι, δηλαδή αντιδρούμε ως νομοθετικό ε, σώμα το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μαζί. Καλή εξέλιξη αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μία αποδεκτή λύση για όλα τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα εργαλεία που διαθέτουμε όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας. Την επόμενη φορά που θα έρθω θα έχω να σας πω περισσότερα γι' αυτά. Τώρα, ποιες είναι οι προοπτικές μετά μετά την επόμενη εβδομάδα. Για, μετά το τρίτο κεφάλαιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα έχουμε ένα σχέδιο κειμένου για τα νομοθετικά μέσα που είναι το 4, το 5 που θα είναι κατεξοδότηση και πράξεις, το 6 που θα είναι ο συντονισμός της νομοθετικής διαδικασίας, 7 ένα ενδιαφέρον θέμα εδώ είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, τη θέση σε ισχύ. Συγκριτικοί πίνακες, κάτι σας λένε αυτά. Κεφάλαιο 8, απλοποίηση και κεφάλαιο 9, εφαρμογή και έλεγχος της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών. Η συμφωνία αυτή για μας μπορεί να αντικαταστήσει την προηγούμενη, αλλά όχι τη συμφωνία πλαίσιο του 2010. Η πρόταση λοιπόν είναι ότι για τα κεφάλαια 4 έως 9 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα βάλουν στο τραπέζι συγκεκριμένα κείμενα ώστε να μπορέσουμε αμέσως να δούμε πού παραμένει πρόβλημα μεταξύ των τριών οργάνων. Το Συμβούλιο ζήτησε για το 5 όσον αφορά τις κατεξουσιδότητες και τις εφαρμοστικές πράξεις που είναι επίμαχο το κεφάλαιο αυτό να συζητηθεί χωριστά από τα υπόλοιπα κεφάλαια. Πάντα είναι επικίνδυνο να προσπαθεί κανείς να προβλέψει το μέλλον, πόσο μάλλον στην πολιτική και γνωρίζουμε ότι τρεις μήνες στην πολιτική είναι μια αιωνιότητα. Όμως πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε επιτυχώς μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και πιστεύω επίσης ότι με τέτοιες συζητήσεις μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ οι σχέσεις μεταξύ των τριών οργάνων. και είναι πολύ καλό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να δούμε το κλασικό νομοθετικό έργο και να προχωρήσουμε βάσει αυτού, δηλαδή πρώτα διαβούλευση, μετά πρόταση. Ολοκληρώνω εδώ. Όταν για τα κεφάλαια 3 και 4 θα έχουμε συμφωνία, προτείνω να επανέλθω για να σας ενημερώσω και πάλι για το που βρισκόμαστε και για να απαντήσω και σε ό,τι ερωτήσεις θα έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση. Λοιπόν, η Σιλβί Κάφμαν πρώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα Γκί για τις πληροφορίες και εύχομαι καλή τύχη και να τα καταφέρεις να ολοκληρώσει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Κάτι πραγματάκια θα ήθελα να αναφέρω που θα ήθελα να ενισχύσω την θέση του Γκίφερ Χόφστατ. Το ένα είναι το θέμα της απόσυρσης προτάσεων. Έχουμε ζήσει το ότι η Κομισιόν απέσυρε κείμενα τα οποία είχαν προχωρήσει πολύ στο Κοινοβούλιο, είχαν περάσει την πρώτη ανάγνωση και μετά τα απέσυρε Κομισιόν με το επιχείρημα ότι δεν, υπήρχε, δεν προβλέπεται να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο. Πολιτικά δύσκολο Ξέρουμε πως είναι η κατάσταση, υπάρχει ακόμα και απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν ξέρω γιατί η Κομισιόν συμπεριφέρεται διαφορετικά στον έναν από τους δύο νομοθέτες. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην ε, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χρειάστηκαν μέχρι και 20 χρόνια για να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μας λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, ότι θα χρειαστούν τέσσερα χρόνια ξέρω εγώ και δεν έχει άρα σημασία το τι λέει το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Και θεωρώ πως εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στην Κομισιόν, να απαιτήσουμε από την Κομισιόν ίση μεταχείριση των δύο συνομοθετών. Το δεύτερο, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι το θέμα της αξιολόγησης ε, αντικτύπου. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το πρόγραμμα REFIT ε, και όπως και να έχουν τα πράγματα θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό και το είπα κιόλας ε, πως όταν γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν μόνα τους όταν εμείς θεωρούμε ως κοινοβούλιο ότι κάνουμε σοβαρές προτάσεις αλλαγής μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε το τι θα γίνει με την αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συστήματα αξιολόγησης αντικτύπου όπου θα κάνουν την αξιολόγηση αυτοί που θα αφαιρούν μετά το δικαίωμα του νομοθέτη να λάβει πολιτικές αποφάσεις. Εντάξει, υπερβάλλω, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια τάση τέτοια από πλευρά ε, κομισιών. Μιλάει εδώ πέρα για έναν εξάρτητο πάνελ, ποιοι θα είναι αυτοί. Ε, είναι πάρα πολύ προβληματική η κατάσταση και δεν είναι δυνατόν να την δεχτεί το Κοινοβούλιο. Ε, μπορούσα να πω και άλλα πολλά αλλά θα μείνω σε αυτά και εύχομαι καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, Ράμαν Χάουρικ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τον Κι για τις ε, πληροφορίες και να του υποβάλω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο ερώτημα είναι δεν ξέρω αν κατά πόσο σε πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτό θα εξεταστεί και η παρακολούθηση ή συνέχεια σε νομοθετικές πρωτοβουλίες πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλώ για εκθέσει πρωτοβουλία. Το Κοινοβούλιο εγκρίνει γύρω στις 50 εκθέσεις πρωτοβουλία κάθε χρόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως η Κομισιόν είναι κάποια συνέχεια. Αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός δηλαδή που θα μελετά τι αντίκτυπο έχουν οι εκθέσει πρωτοβουλία μα ε, στο έργο τη Κομισιόν. Δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται στην εντολή του Γκί. Θα ήθελα να μου πει πάντω. Γιατί πράγματι με απασχολεί το κατά πόσον οι εκθέσει μα μπαίνουν σε ένα σιρτάρι ή κάτι κάνουν τελικά, κάποια χρησιμότητα έχουν. Δεύτερο ερώτημα. Το σχέδιο Τίμπερμανς, ο αντιπρόεδρος μας παρουσίασε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης όλων των προτάσεων, οδηγιών, κανονισμών που συζητούνταν ε, σε επίπεδο Κομισιών και Συμβουλίου. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να δίνει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να δει τι θα αποσυρθεί, τι δεν θα αποσυρθεί, υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου αυτού του σχεδίου του Αντιπρόεδρου της Κομισιόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Γκερέρο Σάλομ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον Γκί για τις πληροφορίες που μας έδωσε σε σχέση με την πρόοδο αυτών των διαπραγματεύσεων που ελπίζουμε να ολοκληρώσουν, να ολοκληρωθούν συγγνώμη, σε εύθετο χρόνο. Γιατί είπα ότι τρεις μήνες στην πολιτική είναι μια αιωνιότητα. Ξέρετε όμως πολλές φορές ε, τρεις μήνες τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι τίποτα. Τίθεται ένα θέμα, πάμε σε μια συνεδρίαση, ξανατίθεται το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, μετά εγκρίνεται ότι θα παραπευθεί η εξέταση του θέματος σε μια προσεχή συνεδρίαση, μετά υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία που τίθεται υποσυζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση και ούτω καθεξής. Και λίγο να μην προσέξουμε έχει περάσει μισή χρονιά ή μισή νομοθετική περίοδος θα έλεγα ακόμα καλύτερα και μετά μας παίζει ο χρόνος. Φαντάζομαι, νομίζω ότι συμφωνεί και ο Γκί, ε, ότι καταλαβαίνει και αυτός ότι είναι ανάγκη να επιταχύνουμε και να καταλήξουμε ή δυνατόν βέβαια στη συμφωνία αυτή. Εμένα μου δίνεται η εντύπωση ότι δεν θα υπάρξουν ε, σοβαρά προβλήματα στο κεφάλαιο προγραμματισμός Νομίζω ότι είναι λογικό τα κεντρικά ε, σημεία της νομοθεσίας να αφορούν τη συζήτηση, ε, τις προγραμματικές δηλώσεις ουσιαστικά, το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Κομισιόν, κατάσταση της Ένωσης και επίσης παρουσία του Συμβουλίου, γιατί αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Παρουσία του Συμβουλίου για κάθε θέμα που συζητείται και αφορά την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Αυτό το θέαμα να λαμβάνονται αποφάσεις στο Κοινοβούλιο για πολύ σημαντικά ζητήματα στο ε, πλαίσιο της κοινοβουλευτικής περίοδου με άδεια τα έδρανα ε, του Συμβουλίου νομίζω ότι δεν περιπεί και πρέπει και το Συμβούλιο να συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις θεμελιώδεις συζητήσεις που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όχι μόνο όταν πρόκειται για συνεδρία του Συμβουλίου, αλλά γενικά για τι δραστηριότητε των θεσμικών οργάνων. Επίση, όπω είπε η σύντροφο Κάφμαν, και εν μέρει νομίζω είπε και ο κ. Φερχόφστατ, ότι θα υπάρξουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τι εξολογήσει αντικτύπου. Θα υπάρξουν προβλήματα ως προς το περιεχόμενο και ως προς το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, όπως ε, προδιαγράφεται το σενάριο αυτή τη στιγμή, να γίνει μια εκ των υστέρων, εξολόγηση να υπάρχει και μια εκ των προτέρων, αξιολόγηση με συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, μετά με διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους και ούτω καθεξής, τελικά δίνεται ενδεχομένως η εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας ακρίκος απλά μέσα σε όλη αυτή την ε, νομοθετική διαδικασία. Ο κύριος Τίμερμανς πράγματι επανειλημμένος έχει πει ότι η τελική πολιτική απόφαση είναι ε, στο κοινοβούλιο. Επομένως, οι αξιολογήσεις, αν έχουν κάποια χρησιμότητα, αυτή είναι για να δώσουν ε, μια καλύτερη εικόνα ε, στο κοινοβούλιο και να τους δώσουν τις πληροφορίες ώστε να μπορέσει να πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Αν όμως στο τέλος προκύψει ότι έχουμε πληθώρα ε, φορέων όπου εκεί η πολιτική απόφαση συγχέεται με την τεχνική αξιολόγηση, την εξωτερική συμμετοχή και άλλους φορείς που αντιπροσωπεύουν εθνικές κυριαρχίες όπως τα εθνικά κοινοβούλια, τότε ε, θα υπάρξει μια περίοδος σύγχυσης. Το έχω πει ε, σε άλλους, δεν ξέρω ε, αν το έχει ακούσει ο κ. Φερχόφστα, το φιλόσοφος Μπέικον είχε πει ότι περισσότερο πιθανότητε είναι το σωστό να προκύψει από το λάθος παρά τη σύγχυση. Άρα μέσα στη σύγχυση πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες να κάνουμε λάθος. Είναι πολύ σημαντικό όμως και το περιεχόμενο, δηλαδή αξιολόγηση, να μην είναι μια αξιολόγηση κόστους ωφέλους, αλλά να λαμβάνει υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, περιβαλλοντικά κριτήρια. Να είναι μια κοινωνικά υπεύθυνη αξιολόγηση να μην ε, βλέπει μόνο τα κέρδη και τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν από έναν κανονισμό. Επίσης, ε, όπως είπε και ο κύριος ε, Φερχόφστατ, πράγματι τίποτα δεν, είναι, δεν έχει συμφωνηθεί αν δεν συμφωνηθούν όλα, τα πάντα. Το θέμα είναι βέβαια να παραβιάζονται κάποιοι κανόνες της διαπραγμάτευσης. Αν όμως υπάρχει συμφωνία για συγκεκριμένα κείμενα, καλό θα ήταν η Επιτροπή Αύκο να λαμβάνει γνώση των κειμένων αυτών. Επαναλαμβάνω, αν δεν παραβιάζονται κανόνες της διαπραγμάτευσης, για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο τη διαδικασίας. Αρκεί, όπως είπα, να υπάρχει ένα επίπεδο συμφωνίας που να αφήνει να εννοηθεί ότι θα υπάρξει τελικά συμφωνία. Παραλαμβάνω μπορούμε να ελέγχουμε για να βλέπουμε αν πηγαίνει το πράγμα ε, όπως επιθυμεί το Κοινοβούλιο. Ο κύριος ε, Σταχόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο ήταν ε, ενδιαφέρον για μένα ήταν ένα κομμάτι αυτών των οποίων είπατε και σας ευχαριστώ κύριε Φερχόφτα που ήρθατε και μας παρουσιάσατε αυτή την έκθεση ήταν το κομμάτι που είπατε ότι υπάρχει μια κάποια σύγκρουση μεταξύ αξιολόγησης αντικτύπου όταν μιλάμε για τροπολογίες που υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην νομοθετική διαδικασία. Οπότε αφενός αυτό μπορεί να το δει κανείς ως μια προσπάθεια να περιοριστούν οι νομοθετικές αρμοδιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αλλά ίσως υπάρχει και κάποια ουσία εδώ πέρα. Ξέρουμε πως 80% των, ε, της νομοθεσίας εγκρίνεται στην πρώτη ανάγνωση. Έχουμε μια ιδιαίτερη νομοθετική διαδικασία, οπότε κάποιο βήμα προς τα εμπρός, ε, προς την πρόταση της ε, Κομισιόν, ίσως να είναι θετικό, γιατί γεγονό είναι πως η καλύτερη ρύθμιση και η νομοθεσία είναι ο κοινό μας στόχος. Δεν είναι μόνο θέμα σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η άποψή μου λοιπόν θα δούμε τις δικές μας και το τι μπορεί να αλλάξει εκεί πέρα και ίσως ε, λιγότερες τροπολογίες αλλά πιο ουσιαστικές. Για να δούμε το τι θα γίνει με την ουσία του κάθε θέματος. Βεβαίως υπάρχουν συχνά οι φόβοι ότι προσπαθούν εδώ πέρα να περιορίσουν τις νομοθετικές μας ε, αρμοδιότητες. Και βεβαίως κύριε Φερχόφστατ, εσείς με την πείρα σας ε, έχετε μια καλή εικόνα για το τι γίνεται σε σχέση με τον ρόλο των θεσμικών οργάνων. Οπότε θα έπρεπε νομίζω ίσως να δούμε το τι κάνουμε και να δείξουμε λίγη ευαισθησία και νομίζω καλύτερη ρύθμιση θα σημάνει λιγότερη γραφειοκρατία. Παραδείγματο χάρη στον τριμερή διάλογο κάθε μέρος θα πρέπει να έχει δυνατότητα να επανέλθει με ερωτήσεις ε, ε, στη διάρκεια της ε, αξιολόγησης αντικτύπου. Όχι σε κάθε τροπολογία, εντάξει, γιατί θα διαλυθεί η διαδικασία, αλλά ίσως για κάποιες ε, τροπολογίες κλειδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις. Η μία αφορά τα εθνικά κοινοβούλια και τον ρόλο τους στην ευρωπαϊκή λήψη αποφάσεων. Θεωρείτε πως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μπορούν να εμπλακούν στη διαδικασία και να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για τον ρόλο τους. Μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τις διάφορες ε, διαβουλεύσεις. Γιατί κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ε, διαδικασία. Και προσωπικά πιστεύω πως ε, είναι σημαντικό η Κομισιόν να συνεχίσει την ε, διαδικασία αυτή ε, για να μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εκφράζονται, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου θα διαβουλευόμαστε επί νομοθετήματος που έχει ήδη εγκριθεί. Πριν λοιπόν η Κομισιόν λάβει μια τελική απόφαση, όταν είναι έτοιμη όμως η πρότασή της, εκεί πέρα νομίζω μπορεί να γίνει η πραγματική διαβούλευση. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Μπορούμε να έχουμε μια αρχική περίοδο διαβούλευσης με την ε, πράσινη βιβλό. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν ε, άλλες ε, ερωτήσεις από τους συναδέλφους θα δώσω τον λόγο στον Κίφερ Χόφστατ. Χωρίς μικρόφωνο, κύριο Χόφστατ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνοψίσω κάποια πραγματάκια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα για τον προγραμματισμό, το πρόβλημα της απόσυρσης ε, που αναφέρατε. Πράγματι προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ίση μεταχείριση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γιατί υπάρχει πίεση του Συμβουλίου από καιρού εις καιρών, αλλά νομίζω πως ακολουθούμε εδώ πέρα περισσότερο τις επιλογές και τις επιθυμίες του Συμβουλίου και όχι τόσο του Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια ίση μεταχείριση. Δεν μπορούμε τώρα να προβλέψουμε κάποιες διαδικασίες γι' αυτό, απλά θα πρέπει να φροντίσουμε ότι ε, και στα αιτήματα πρωτοβουλίας προς την Κομισιόν και στα αιτήματα απόσυρσης ενός φακέλου Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να είναι απολύτως στο ίδιο επίπεδο. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε τις, το μέγιστο αριθμό εγγυήσεων. 100% βεβαίως αυτό δεν γίνεται. Οπότε α, δεν ξέρω αλλά θα πρέπει να τους ε, το επιβάλλουμε γιατί να έχουν την ίδια αντίδραση δηλαδή όταν ζητάει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μια πρωτοβουλία. Αλλά κοιτάξτε, αυτό υπάρχει ε, ούτως ή άλλως το κείμενο ως ίση μεταχείριση. Επίσης, ε, στην έκθεση Δίας Πρωτοβουλίας, τι είναι αυτό, είναι κατ' ουσίαν ένα αίτημα προς την Κομισιόν για να κινητοποιηθεί, για να καταθέσει μια νομοθετική πρωτοβουλία. Ίσως ε, να μην έχουν ούτε μία σχέση με την Κομισιόν, αλλά όταν μιλάμε για μια εκθέση δύο που ζητάει κάτι από την Κομισιόν, είτε πρόκειται για δράση είτε για νομοθεσία, τότε νομίζω πως καλύπτεται από τις διατάξεις που έχουμε τώρα. Αλλά βεβαίω ε, δεν έχουμε ποτέ 100% εγγύηση ίσης μεταχείρισης ε, γιατί εξαρτάται και από το πώς εργάζεται η Κομισιόν. Τώρα για την αξιολόγηση αντικτύπου για αυτά τα οποία είπε η κυρία Κάφμαν για την έκθεση Ρίφιτ. Να ξεκαθαρίσω λίγο κάτι το εξή. Το πώς το βλέπω εγώ. Εγώ ποτέ δεν θα αρνηθώ το να κάνει μια αξιολόγηση αντικτύπου ένα θεσμικό όργανο. Αν θέλει να κάνει η Κομισιόν ε, μια αξιολόγηση αντικτύπου σε δική της πρόταση ή σε τροπολογία του Κοινοβουλίου του Συμβουλίου είναι δικαίωμα της, όπως είναι και δικό μας άλλωστε. Αυτές νομίζω ότι είναι οι βασικές αρχές. Η βασική αρχή είναι όμως ότι δεν μπορούμε να τα αναθέσουμε αυτά σε οποιονδήποτε, στον οποιονδήποτε. Όχι. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε κάποιον εξωτερικό, ούτε η Κομισιόν, ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν έχω λοιπόν τίποτα με την αξιολόγηση αντικτύπου. Απλά λέω πως δεν μπορούμε να το αναθέσουμε σε τρίτο και να λέμε «Α, ναι, τώρα η Κομισιόν θα τα κάνει και εμείς δεν μας δεσμεύει» κτλ. Όχι, δεν πάει έτσι. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να κάνουμε δική μας αξιολόγηση αντικτύπου, να πούμε πως εντάξει, μια αξιολόγηση αντικτύπου που έκανε η Κομισιόν είναι καλή και τη λαμβάνουμε υπόψη, αλλά μπορεί και μια αξιολόγηση αντικτύπου ακόμα και σε έναν τριμερή διάλογο μπορούμε να μπορούμε για να ξεφύγουμε από ένα αδιέξοδο να κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Αλλά η αρχή δεν είναι να είμαστε κατά των αξιολογήσεων αντικτύπου, αλλά να μην παραδώσουμε την νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου όπως δεν το κάνει ούτε το Συμβούλιο. Αν μας πούνε δηλαδή ότι κάναμε μια αξιολόγηση αντικτύπου και τώρα θα την ακολουθήσουν όλοι γιατί είναι αντικειμενική. Ε, όχι, συγγνώμη, τι θα πει αντικειμενική δηλαδή τη σήμερον ημέρα. Ούτε και οι εκπομπέ των αυτοκινήτων πλέον δεν είναι τόσο αντικειμενικές. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι το αντικειμενικό, αλλά προφανώς δεν είναι. Λοιπόν, μην με παρεξηγείτε, το πρόβλημα δεν είναι ε, ναι ή όχι στην αξιολόγηση αντικτύπου, είναι ποιος την κάνει και τι συνέπειες έχει. Και ναι, εγώ είμαι υπέρ, αλλά και νομίζω πως και το Κοινοβούλιο Μπορεί να, αλλά να δεχτούμε την απόφαση Κομισιόν ή να την απορρίψουμε, αλλά είναι δικό μας ε, το προνόμιο να διαλέξουμε έτσι και μπορεί να λαμβάνουμε διαφορετική απόφαση κάθε φορά. Μπορεί, κάθε φορά να, ε, μπορεί μια φορά να πούμε ότι καλύτερα να κάνουμε μία αξιολόγηση αντικτύπου ή το αντίστροφο. Αλλά θα το ε, αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν ότι η αξιολόγηση αντικτύπου που κάνει ένα θεσμικό όργανο είναι και η επίσημη αλήθεια και εκδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Θα προβλέπονται βεβαίως ε, αξιολογήσεις αντικτύπου. Ε, μπορεί να γίνουν διάφορες φάσεις, ε, αλλά ακόμα και σε έναν τριμερή διάλογο, αλλά τότε πρέπει όλοι να συμμετέχουν. και δεν είναι δυνατόν να τις κάνει μόνο ένα θεσμικό όργανο. Μετά, για τα εθνικά κοινοβούλια. Κοιτάξτε, αν υπάρχει η δυνατότητα, μιλήσαμε για τον τριμερή διάλογο, διαφάνεια κτλ. Ίσως να το δούμε αυτό αναλόγως ε, το κλίμα ε, γύρω από το τραπέζι, για τα εθνικά κοινοβούλια εδώ πέρα ε, καθορίζει μια διαδικασία ή συνθήκη. Η κόκκινη κάρτα, η κίτρινη κάρτα και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. εντάξει να το κάνουμε, αλλά στο πλαίσιο που υπάρχει, έτσι. Τούτου λεχθέντος βεβαίως είναι ένα ζήτημα οπωσδήποτε το οποίο θα είναι επιτάπητος ε, και στην ε, έκθεση προόδου και ίσως και στη δική μου έκθεση. Αλλά αυτό το οποίο εγώ θεωρώ είναι πως ε, το εθνικό, το ευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχει το ευρωπαϊκό επίπεδο και τα εθνικά κοινοβούλια ελέγχουν το εθνικό επίπεδο και καλό είναι να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το να τα ανακατεύουμε όλα, ξεχάστε το. Δεν υπάρχουν αυτά που θένα. Και ειδικά αυτές οι ιδέες ε, που ακούω που λένε ναι έχουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες και το Συμβούλιο εκπροσωπεί τα κρατημέλη και χρειαζόμαστε ένα τρίτο ε, κομμάτι με εθνικά και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Μα ξεχάστε τα, εμείς τι θα είμαστε, η μόνη δημοκρατία στον κόσμο με τρία κοινοβουλία. Δεν θα πάω σε αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι για το θέμα της διοργανικής ε, συμφωνίας, αλλά δεν μπορεί να τα ανακατεύουμε τόσο πολύ. Να ξεκαθαρίσουμε τι κάνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Το να τα ανακατέψουμε, όχι. Δεν ε, θέλω εγώ τουλάχιστον να πάρω τι διαπραγματεύσει. Επ' αυτού. Νομίζω ότι θα το κάνετε γιατί όντω πρέπει να έχουμε γραπτά αυτή την προσέγγιση. Γιατί νομίζω ότι θα συνεχίσετε να έχετε διαφωνήσει και πολλά προβλήματα για να υπάρχει μια κοινή κατανόηση και κοινή προσέγγιση από όλα τα όργανα. Θα έχω αυτά αν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει η ευκαιρία να διευκρινιστούν οι ρόλοι, φυσικά και πρέπει να το κάνουμε. Σίγουρα, φόσον και τα τρία όργανα έχουν την ίδια απόψη. Ωραία. Λοιπόν, Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ελπίζω Μόλις έχετε κάτι καινούριο, να επανέλθετε. Και είστε πάντα ευπρόσδεκτος και σε κάθε συνεδρίασή μας, άμα θέλετε, να μας το πείτε από πριν. Και ελπίζω, άμα θέλετε να τελειώσετε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ωραία, έληξε η συνεδρίαση τον Οκτώβριο και πάλι θα συνεδριάσουμε.